Ζητώ συγγνώμη για την τετράλεπτη καθυστέρηση. Α, δεν βλέπω και το ρολόι. Δεν έχουμε ρολόι. Α, δεν το βλέπω από εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Ε, ε, θα μπλέκουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είναι στο πλάι τα ρολόγια, γι' αυτό δεν τα βλέπετε. Είναι πίσω από την πλάτη μου. Ωραία, να μου λέτε τότε πότε να σταματάω. Είναι φορτωμένη η μερίσια διάταξη σήμερα. Θα προσπαθήσουμε ε, να ε, εξαντλήσουμε το πρόγραμμά μας και χρονικά έγκριση μερίσια διάταξης. Θα πρότεινα να ε, κάνουμε δύο λαγέ στο σχέδιο μερίσια διάταξης. Ελπίζω να σας τα έχουν πει αυτά οι σύμβολοι των πολιτικών ομάδων, γιατί και εμένα οι σύμβολοι μου τα λένε και η γραμματεία, λόγω της τεχνικής πελιπλοκότητας και των πολιτικών δυσκολιών, προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για δύο θέματα, InvestEU, με εισηγήτρια την κυρία Βέστφαλ και η διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη ε, με εισηγητή τον κύριο Πιτρόφσκι. Επειδή οι αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές έχουν επίσης αναβάλει ε, τη συζήτηση και το χρονοδιάγραμμά τους, μπορούμε να τα ψηφίσουμε τα θέματα αυτά εν ευθέτω χρόνο όντας πάντα εμπρόθεσμοι για τις επιτροπές που γνωμοδοτούμε. Αν συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερησία διαταξή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω καμία ανακοίνωση να σας κάνω, διότι χρειαζόμαστε πολύ χρόνο για την ψηφοφορία. Και αρχίζουμε τώρα αμέσως με τις ψηφοφορίες πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ε, ιδρύοντας το Ορίζον ε, Ευρώπη, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία καθορίζει ε, τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης. Είναι του κυρίου Βανίστερ η γνωμοδότηση. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς τα είπατε κι εσείς ότι πρέπει να επιταχύνουμε. Ε, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή έχει πατήσει γκάζι, δεν σταμάτητη είναι. Και θα πρέπει να εγκρίνουμε εμείς την γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης και την ε, γραμματεία. Ήταν πολύ καλή υποστήριξη και προχωρήσαμε δουργά ε, Και τηρήσαμε και τις διατυπώσεις του Γενικού Κανονισμού για τις άμεσες ε, μεταφορές ε, σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό. Συμφωνήσαμε για κάποιες τροπολογίες και νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσω στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί ομαλά κατά την άποψή μου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ε, μπορούμε λοιπόν να περάσουμε αμέσω στην ψηφοφορία. Στο συγγνώμη, έχω προβλήματα εδώ <laughs> με τα μηχανήματα, με το... Δεν ξέρω. Εσείς ε, υπάρχει κάποιος τεχνικός να με βοηθήσει. Δεν δουλεύει το μηχάνημά μου. To, It is not with the card. It is with with device. Ah, yes. Δεν φταίει η κάρτα, λέει η πρόεδρος. Φταίει το μηχάνημα. Λοιπόν, προχωρούμε. Ζητώ συγγνώμη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε μαζί τροπολογίες 147, 148, 187, 249 και 125. Όλες αυτές μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Μπορούμε παρακαλώ να το επαληθεύσουμε για καλό και για κακό. Δουλεύουν όλα τα μηχανήματα ή κανένα. The vote is open. No. Αρχίζει η ψηφοφορία, θεωρητικά. Α, τώρα άνοιξε. Αυτό ήταν το Σουσάμι άνοιξε, έπρεπε να πω αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Hey. <laughs> yes, please. Η κυρία Εράτσε Γκαρθία να μετρηθεί η ψήφος μου. Δεν ψήφισα, μου φέρνουν τώρα το, την ε, κάρτα μου που την έχω ξεχάσει στην Ολομέλεια. Είμαι από την αρχή εδώ της συνεδρίασης, απλώς δεν είχα την κάρτα μου. Παρακαλώ αν καταγραφεί η ψήφος μου. Μπορείτε να επαναλάβετε, λέει πρόεδρος. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχω την κάρτα μου. Είμαι εδώ από την αρχή της συνεδρίασης. Μου τη φέρνουν τώρα, είναι στην Ολομέλεια η κάρτα μου. Τουλάχιστον σηκώνει το χέρι να λες πώς ψηφίζεις. Υπέρ κατά. Λοιπόν, είστε υπέρ. Δεν γκρίνεται λοιπόν. You have today the golden finger. Εσείς είστε οι χρυσοδάκτυλοι σήμερα. Χρυσή ψήφος. Προχωρούμε. Συμβιβασμός υπάρχει 21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Προχωρούμε σε επόμενη συμβιβαστική 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Ε, 23 is in favor. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 188. Ψήφι υπέρ. 188. Και τι γίνεται με την 147, ρωτάει κάποιος. Μα ήταν στο πρώτο μπλοκ που ψηφίσαμε. Προχωρούμε στη συμβαστική 24, γιατί 188 καταπίπτει και αυτή. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμή 25. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα πρέπει να πάμε στη συμβαστική 27, αλλά σας συνιστώ να ψηφίσουμε πρώτα την τροπολογία 234. 224, συγγνώμη, συμφωνεί ο εισηγητής. Για λόγους ε, ευ... δεν διαφωνώ αλλά ε, προτείνω να την καταψηφίσουμε. Αν ψηφίσουμε πρώτα τη 2.34, ε, κατά προτείνω. Ευχαριστούμε για τη συμβουλή. Ωραία. Ψηφίζουμε πρώτα την 2.34. Ψήφι Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τσεκ. Ας το ελέγξουμε λοιπόν. 234. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιατί ψηφίζω και εγώ κατά. Που δεν δουλεύει η κάρτα μου εδώ. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Δεν έχετε το αποτέλεσμα. 15 υπέρ, 18 κατά και μία αποχή. Εντάξει. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε στη συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 250 τώρα. Ψήφι περ Κατά. Αποχές απορρίψεται. τροπολογία 251. Ψήφι περ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 252. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 254 όχι ε, ε, καταπεπτεί 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 31 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 200. Ορίστε. Η κυρία Κρέλ, πρέπει να ανακοινώσω ότι οι τροπολογίες 262, 265, 231 και 141 αποσύρονται. Είναι και σε πακέτα συμβιβασμών. Ωραία. Ε, έχουν αποσυρθεί αυτές. Σας ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Άρα θα προχωρήσουμε στην 267, η οποία δεν έχει αποσυρθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί. 271 υπέρ κατά αποχές, ας το ελέγξουμε αυτό, είναι η τροπολογία 271 παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται λέει η πρόεδρος. Λέει 18-14. Uh, yes, it is, it is... Α, δηλαδή εγκρίνεται. δεν το υπολόγισα σωστά, εγκρίνεται. 272. Ορίστε. Η κυρία Κρέλ. Αυτή η τροπολογία εντάσσεται στο συμβιβασμό υπαριθμών 18 ε, που ψηφίσαμε προηγουμένως ή που θα ψηφίσουμε αργότερα. Αν εγκριθεί η συμβαστική 18 η τροπολογία 272 καλύπτεται από το Συμβασμό 18 που, δεν... που... ψηφίστηκε λέει η Πρόεδρος και εγκρίθηκε. Πάμε στη 273. Συμφωνείτε. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 277. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 288 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 35 με την προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανεί με την προφορική που βλέπετε στον κατάλογο. Όχι, μαζί με την τροπολογία αυτή η 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα περάσουμε στην τροπολογία 291. Ψήφι υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 292 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παρήθμη 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 315 γράφει εδώ. Ναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 63 υπέρ. Α, έχει αποσυρθεί, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 71 η οποία ταυτίζεται με την 72, όχι, όχι, 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Είναι ταυτόσιμη με την 73, ζητώ συγγνώμη. Οπότε τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ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 Η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 110 ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 ε, συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 121 έχει αποσυρθεί. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 130 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 141, συγγνώμη έχει αποσυρθεί και πάμε τώρα στη συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε αυτής. «35 υπέρ» και εγώ μαζί «36». Και εσείς κυρία Γκαρθία ήρθε η κάρτα σας. Όχι, όχι, 36, έχει έρθει η κάρτα. Και ο κύριος Κοτσολίνο, 37, 38. Όχι, εγώ έχω κάρτα, λέει η κυρία Γκαρθία. Ωραία, 37. Ναι, γιατί δική μου δεν λειτουργεί, λέει η πρόεδρος ακόμα. Λοιπόν, 37 υπέρ. Ε, μία ψήφος ε, κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Βανίστελ Ρόι. Και πρέπει να πω και συγχαρητήρια σε όλους μας, γιατί ήταν το πρώτο νομοθετικό θέμα που ψηφίζουμε ε, με το νέο πλαίσιο. Και πολύ μεγάλη επιτυχία και μπράβο μας. And we now τώρα με ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε την κυρία Μπρέζο Γνωμοδότη Επιτροπή Ρέτζη για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Θέλετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να πω και εγώ λίγα λόγια. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την δουλειά, τη γρήγορη δουλειά που κάναμε στο θέμα αυτό. Θεωρώ ότι οι συμβιβαστικές ε, προτάσεις ανταποκρίνονται στο κοινό αίσθημα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να παραμείνει πυλώνας ε, της πολιτικής συνοχής. Αυτή είναι η ουσία των συμβαστικών τροπολογιών και θα έλεγα ότι εργαστήκαμε με τρόπο ώστε να λαμβάνει όσο δυνατόν ε, υπόψη τις απόψεις όλων των συναδέλφων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να το δούμε αυτό στην ψηφοφορία. Ναι. Ευχαριστώ. Περνάμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες. Ε, ξεκινάμε με την τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 107 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Εγώ είμαι κατά όμως, λέει η πρόεδρος. 19-19. Α, και εσείς είστε υπέρ. Α, δουλεύει. 19-19 καταπίπτει. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν 111 με προφορική τροπολογία. Είναι κάποιο κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι, ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά ας τη δούμε 112 λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε. Απορρίφθηκε με την δική μου την ψήφο. Ναι. Ε, καταψηφίσατε δηλαδή, μάλιστα. Ωραία. Απορρίπτεται λοιπόν. Οπότε... 113. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Το ίδιο. Το ίδιο. Θέλετε να το επαληθεύσουμε. Όχι. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία. 113. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ετελείωσε. Και απορρίπτεται. Το ίδιο. Το ίδιο αποτέλεσμα. Συμβαστική ένα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δύο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 με προφορική τροπολογία. Κατά της προφορικής τροπολογίας όχι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία. Συμβιβαστική όχι. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ, όχι. Ναι. Νομίζω όλοι ξέρουν ότι είναι εκείνη η αρμοδιότητα με την Επιτροπή Απασχόλησης και Περιβάλλοντος. Ναι. 148 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 149. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141 ε, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά να σας παρακαλέσω να σηκώσετε το χέρι σας υπέρ την 155 υπέρ κατά αποχές να το δούμε να το επαληθεύσουμε δεν ε, με βοήθησε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ναι, το ψηφίσαμε. Ναι, 157 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 186 καταπίπτει. Όχι, ναι. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να το επαληθεύσουμε μάλιστα. 187 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 188 καταπίπτει γιατί έχει εγκριθεί 87 και περνάμε τώρα στην 190 91 και 92 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 15 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί αν θέλετε μπορούμε να το δούμε εγκρίνεται 209. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 200 13. Ναι, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 221 καταπίπτει. Ναι. 214. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει σχεδόν ταυτόσημη. Ο λίγο έγκυος δηλαδή. Τι είναι αυτά να το ψηφίσουμε χωριστά γιατί είναι σχεδόν ταυτόσιμες. 214 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ. 26 υπέρ. Δεν είναι σχεδόν ταυτόσιμες. Σχεδόν ψηφίζουμε. Ε, από το περιεχόμενο καταπίπτει. Μου λένε εδώ πέρα εγκρίνεται σχεδόν. Σχεδόν συμφωνείτε, όχι. 215. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 216 καταπίπτει. Και περνάμε συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, καταπίπτει, α, συγγνώμη. και καταπίπτει και τώρα έχουμε την 2.27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 231 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 232 ταυτόσημη με την 31. 233 με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Είναι κάποιος κατά, όχι, ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 240 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 242 υπέρ κατά ναι, όχι, δεν συμφωνείτε. 242 την ψηφίσαμε, εγκρίθηκε, τώρα ψηφίζουμε 243 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 244 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 245 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. 251 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Ε, λόγω της ισοψηφίας απορρίπτεται. 253 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε. 257, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πρώτη, τροπολογία υπερθυμών 1. Άρα όχι, γιατί και εγώ είμαι κατά. Ήταν ε, πλάκα, αλλά σήμερα... Είμαι ένας μεταξύ ίσων, μία μεταξύ ίσων, αλλά τέλος πάντων. Τροπολογία ένα. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Επέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30. Επέρ κατά, αποχές, να ελέγξουμε. 30. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Λυπάμαι πολύ. Όχι ε, για το αποτέλεσμα, για το λάθος μου. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Προφορική. Με την προφορική τροποποίηση της ε, εισηγήτρια υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 65 Επέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με προφορική τροποποίηση, τροπολογία της εισηγήτριας. Για την 65. Εγκρίθηκε με την προφορική τροπολογία. Συμβεστική 28. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73. 73 με προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά της προφορικής. Όχι. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. 73 με προφορική τροποποίηση της εισηγήτριας. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 ψήφοι κατά μαζί με την δική 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, νομίζω. Να ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε για την 74. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρας. Απορρίπτεται. 75. 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή υπέρ. Ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία την 80 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Προφορική 30. Ε, συμβαστική 30, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 31. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 94. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτω. Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγώ ψηφίζω υπέρ, άρα 36 ψήφοι υπέρ, Δύο κατά, δεν αποχαίρει συγχαρητήρια κυρία Μπρέσο. Αυτό ήταν το δεύτερο θέμα που έπρεπε να ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και τώρα συνεχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Ντόιτ, ε, Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι. Ωραία λοιπόν, πάμε απευθεία στις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με την τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80. Σωστά. 80 υπέρ κατά. 80 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102. Ναι, με συγχωρείτε, 100 πρώτα. 100. Πήγα πολύ γρήγορα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. 102. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκατόν εννιά καταπίπτει. 103. 103. Παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104. Καταπίπτει. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παρακαλώ να ελέγξουμε 111 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ναι, 116 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και περάσει και απορρίπτεται. Εντάξει, να τελειώσουμε με αυτήν την ψηφοφορία. Λοιπόν, 116 να την επαληθεύσουμε. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, μπορούμε να ξαναψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εκατόν 1-1-6 6 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και πάλι απορρίπτεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να την παληθεύσουμε. 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. 123 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές η ίδια κατάσταση απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβεβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές Θέλετε να την επαληθεύσουμε. 131. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και κλείνει. Απορρίπτεται γιατί ψηφίζω κι εγώ κατά. Χαίρομαι που, έχω, που είμαι χρυσό δάχτυλος. Ε, συμβαίνει συχνά στα εθνικά κοινοβούλια, το ξέρετε αυτό. Όχι εδώ όμως. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. 132 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 134 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε. 17. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Με τη δική μου αρνητική ψήφο. θα βελτιωθώ. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές να την δούμε 47 ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία και πέρασε και απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές να την δούμε 56. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Και καταπίπτει γιατί καταψηφίζω κι εγώ. Τε, ε, σας υπόσχομαι θα βελτιωθώ στην επόμενη ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, ας ε, την επαναλάβουμε. Είναι η τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη. Η 59 ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και η τροπολογία υπαριθμών 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα θα περάσουμε στην τελική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα και τελειώνει. 36 υπέρ με τη δική μου θετική ψήφο. Είδατε που βελτιώθηκα κι εγώ. Uh, vote in favor. So 36... 36 υπέρ, 2 κατά, χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν, κύριε Ντόιτς. Πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε τώρα με την τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Φίτο. Θέλετε να πείτε τίποτα, κύριε Φίτο. Όχι. Ωραία. Περνάμε μέσω στην ψηφοφορία. Ε, τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, αυτό θέλει έλεγχο μάλλον. Η τροπολογία 2. Ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεν σας έβλεπα. Η τροπολογία 3 καταπίπτει. Και περνάμε στην 4. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 5. Κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 με την προφορική είναι κανείς ε, κατά, όχι, μαζί με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλώς. Και προχωρούμε. Έχουμε και άλλη προφορική τροπολογία νέα παράγραφος 8, όχι 6 διορθώνει πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η νέα προφορική για το νέο κείμενο της παραγραφού 6. Και τώρα πάμε στη συμβαστική 1, ψηφί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Η προφορική και πάλι για το νέο κείμενο που ζητούν σοσιαλιστές υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 με την προφορική. Με την προφορική. Διαφωνεί κανείς με την προφορική. Όχι. 10 με την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε παρακαλώ να το ελέγξουμε αυτό. Δεν χρειάζεται, λέει ο κύριο Βανίστερόι. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά ας το τσεκάρουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Σαφέστατα εγκρίνεται. Η τροπολογία 11 καταπίπτει, διότι εγκρίθηκε η 10. Η τροπολογία 12. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία που αρχίζει. Πέρας. 35 υπέρ. Μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια κύριε Φίτο. Ευχαριστώ πολύ για τις ψηφοφορίες. Very well done. And now... Και πολύ καλά τα πήγαμε. Και πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα, στην ημερήσια διάταξη για σήμερα, που είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Μαρζέ. Αποφάσισε η Ρέτζη να γνωμοδοτήσει προς την Επιτροπή Αλίας για την πρόταση ε, ε, κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου για το Ταμείο Θαλάσσια και Αλίας. Ο κύριος Ομαρζέ είναι συντάκτη γνωμοδότησης που μας παρουσιάζει το σχέδιο της γνωμοδότησής του. Παρακαλώ κάντε λίγη ησυχία στην αίθουσα. Thank you very much. you have the floor. Σας ευχαριστώ πολύ και στο επανειδήν όσοι φεύγετε. Euh, rapidement concernant ε, γρήγορα, ε, Πρόεδρε, για το Ταμείο αυτό της Αλίας είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ταμείο για τη θάλασσα, για την αλία, σημαντικό για τους αλιείς και για όλα τα νησιά, ε, τις παραθαλάσσιες και θαλάσσιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για να προωθήσει τους φιλόδοξους όσο και καινοτόμους στόχους για μια αλία υπεύθυνη και βιώσιμη, για τη διατήρηση των βιολογικών θαλάσσιων πόρων, για την επισητιστική κυριαρχία χάρη ε, στα προϊόντα της θάλασσας, για τη γαλάζια βιώσιμη οικονομία και γενικώ για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστής της διεθνούς ε, ε, διακυβέρνησης και ελέγχου των ωκεανών χάρη στις ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιφέρειες και το λέω από τώρα και στις ε, Υπερπόντιε κτίσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη θαλάσσια δύναμη παγκοσμίω. Το λέμε ξανά και ξανά, αλλά δεν πειράζει να το επαναλαμβάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει ξέχοντα ρόλο εδώ, όσο και ευθύνε ε, σε όλου αυτού του τομεί. Αυτό κάνει η γνωμοδότησή μου και οι προτάσει μου και τα τονίζει όλα αυτά τα θέματα. Η θάλασσα είναι κοινό μας αγαθό, ανεκτήμητο για την ανθρωπότητα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και απολύτως ε, πρωταρχικό είναι να το διατηρήσουμε αυτό το αγαθό και να προσανατολίσουμε τη δράση μας στην προστασία της. Βεβαίως κατανοούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια πολιτική αλίας για τους στόχους αυτούς, τους οικονομικούς και τους αναπτυξιακούς και της περιφερειακής ανάπτυξης. Διότι επιτρέπει να συνδέονται τα διάφορα εδάφη και επικράτειες της Ένωσης και ε, ιδιαίτερα εξόχως απομακρυσμένες. Ξέρετε ότι με την κλιματική απορρίθμιση η βιοπικιλότητα των θαλασσών και των ωκεανών σήμερα απειλείται και επειδή ανεβαίνει η στάθμη των ωκεανών, χρειάζεται σοβαρά να δράσουμε όλοι οι φορείς, οι κοινωνικοί, οι οικονομικοί, οι περιβαλλοντικοί, οι πάντες. Και έτσι λοιπόν, ως πρώτο η Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Επικράτεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κυριαρχεί στην παγκόσμια διακυβέρνηση των ωκεανών, να ενισχύσει τη θέση της και έτσι θα ενισχυθούν και όλα τα ευρωπαϊκά νησιά, όλες οι παραθαλάσσιες περιοχές και το σύνολο ε, των ναυτικών και θαλασσίων περιοχών στην Ένωση. Άρα θα πρέπει ε, να επικεντρωθούμε στη διαφύλαξη των πόρων, στη βιοπικιλότητα, του περιβάλλοντος, πιστεύω το καταλάβατε αυτά. Ε, και θα πρέπει αυτό να μεταφραστεί τουλάχιστον με τη διατήρηση του προϋπολογισμού στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 με ένα ελάχιστο 25% των πόρων που να πηγαίνουν ε, στην προστασία και την ανάκτηση των, ε, της βιοπικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το είχα ξαναπεί την περασμένη φορά για το προηγούμενο Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, την περασμένη θητεία, ότι αν συνεχίσουμε να ρημάζουμε τις θάλασσες όπως το κάνουμε, δεν θα έχουμε ε, κανένα ψάρι ε, όστρακο ή θαλασσινό για την εμπορική αλία πριν το 2050. Η γνωμοδότησή μου που λοιπόν, ανασχολείται με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες και επαναφέρω το σύνολο ε, των ρυθμίσεων του προηγουμένου ταμείου που στη νέα αναθεώρηση έχουν καταργηθεί. Γίνονται και αναφορές στο άρθρο 349 ε, ε, για κάποιες εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 349 για την αλία έτσι ώστε να επανέλθει κάποια ρύθμιση που έχει καταργηθεί. και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην ενδιάμεση ε, αξιολόγηση να κοιτάξει αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα ΠΟΣΕΙ για την αλία δηλαδή ε, που ζητούν όλοι οι βουλευτές των εξόχως απομακρυσμένων περιφερειών. και να έχουν και δραστηριότητα και όχι απλώς να έχουν τη σημαία των από απομακρυσμένων περιοχών και να είναι στον ιολόγιο αυτών των λιμένων χωρίς να έχουν δραστηριότητα εκεί. Επίσης θα πρέπει καλύτερα να προστατεύουμε το περιβάλλον και τη βιοπικιλότητα με χρηματοδότηση δράσεων απορρίπανσης της θάλασσας σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Και από αυτού εχθές, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που αφορούσε τις οδηγίες για τα πλαστικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απορρίπανση των θαλασσών και των ωκεανών. Ε, δική μου τροπολογία που είχα καταθέσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Χρηματοδοτώντας λοιπόν την προστασία των απειλούμενων ειδών, καταπολεμώντας τη λαθρέα αλληλεία και την παράνομη και τη μη δηλωμένη και τη μη ρυθμισμένη, ε, θα ε, βοηθήσουμε και τους ωκεανούς να γλιτώσουν από την επέλαση αυτή του πλαστικού. Επίσης, Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι αλληλείας που δεν είναι επιλέξιμες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, ε, που ρημάζουν τα πάντα, όπως είναι κάποιες στράτες ε, βυθού που τα σαρώνουν όλα ε, και δεν επιτρέπουν την ανανέωση των αλληλευτικών πόρων. Τέλος, σε ό,τι αφορά την διεθνή διακυβέρνηση των θαλασσών και των ωκεανών, κάνω προτάσεις έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κινητήρια δύναμη αυτού του νέου ορίζοντα, ανοίγοντας ε, τα ερευνητικά κονδύλια για την προστασία των μεγάλων θηλαστικών, ε, την απορρίπανση των θαλασσών και τη διακυβέρνηση αυτή καθ' αυτήν. Τούτων όλων λεχθέντων θέλω να πω επίσης ότι όλα τα υπόλοιπα μας βρίσκουν σύμφωνους. Ε, κάνω κάποια σχόλια για όσα πρέπει να αλλάξουν ή να ενισχυθούν. Σε αυτά που συμφωνούμε δεν κάνω καμία αναφορά. Και γενικά θεωρώ ότι η πρόταση είναι ενδιαφέρουσα και ελπίζω να είναι γόνιμη η συνεργασία μας και να μπορέσω να κάνω μια πρόταση ε, φιλόδοξη στην γνωμοδότησή μου για να έχουμε τους στόχους της περιφερειακής ανάπτυξης του Ταμείου αυτού. Thank you. Thank you very Ευχαριστούμε κύριε Μαρζέ και τώρα λόγω στους κοιόδης εξηγητές. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ο κύριος η κυρία Τσουφρίντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα και να παρουσιάσω αυτά που κατά την άποψή μου είναι σημεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση το να επιταχύνουμε και να κάνουμε πιο ε, εύκολες τις διαδικασίες με διοικητικά μέτρα για την πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια είναι ζωτική σημασία. Η αναθεώρηση όμως πρέπει να περιλαμβάνει και στοιχεία ε, καινοτομία για τα προγράμματα. Μεγαλύτερη έλεγχη, περισσότερη έλεγχη, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ε, μείωση του διοικητικού άχθους και του κόστους που, έχουν αυτές για, που έχει αυτό για τις επιχειρήσεις. Χρειάζονται αλλαγές ώστε οι περιφέρειες να, γίνουν, να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο ε, στην εκτέλεση των ε, εφαρμοστικών προγραμμάτων. Αυτό θα επιτρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και με τις τοπικές αρχές και τελικά να ωφεληθούμε οικονομικά, κοινωνικά και ως προς την απασχόληση. Αυτά θα πρέπει να είναι μεταξύ των στόχων μας. Όλα αυτά βεβαίως δεν ε, μπορεί να παραγωνίζει δύο στοιχεία που πρέπει να προβλεφθούν στον μελλοντικό, στο μελλοντικό πλαίσιο προγραμματισμού σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, τουλάχιστον η διατήρηση των ε, πόρων που τώρα προβλέπονται, διότι αυτή τη στιγμή μεταξύ της ε, άμεσης διαχείρισης και της συνδιαχείρισης είναι κάτι που μας ε, κάνει να ανησυχούμε. Θα έχουμε 13% μείωση σε σχέση με τα σήμερα προβλεπόμενα κονδύλια. Η πολιτική αλίας αυτή τη στιγμή βασίζεται στην προσπάθεια μείωσης των αλληλευτικών προσπαθειών για να αποκατασταθούν τα ηθικά αποθέματα. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε όμως την παράκτη αλία, ιδίως την ε, ερασιτεχνική αλία. Ε, και ο κύριος Ομαρζέ θυμίζει, τις, μας μίλησε για τις εξόχως αποκέντρες περιοχές. Όλος όμως ο νότος της Ευρώπης έχει τέτοια μορφολογία και πολύ στενή σχέση ε, και σχέση ζωτική με την αλία την ερασιτεχνική. Θα πρέπει λοιπόν ό,τι μέτρα προβλέψουμε να είναι βιώσιμα και οικονομικά και κοινωνικά. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ήχθιο τουρισμό, τον, την ψυχολογική αλλία, την ε, συγκέντρωση δεδομένων, τη συγκέντρωση πόρων για το μάρκετινγκ των φορέων είναι στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη ο κανονισμός. Κατά δεύτερον, η κατάρτιση και η εκπαίδευση, η ένταξη των νέων σε αυτόν τον τομέα. Εάν θέλουμε να δώσουμε μια όθηση στην αλληλεία του μέλλοντο, πρέπει να μην ξεχνάμε του νέου. Πρέπει να του δώσουμε πόρου για να διαφοροποιηθούν οι δυνατότητε τη ερασιτεχνική αλληλεία. Μάλιστα, διαγράφτηκε από τον προγραμματισμό το τμήμα που αφορούσε την στήριξη των ανθρώπινου κεφαλαίου με τη δημιουργία θέσεων ε, ε, απασχόληση και κοινωνική κοινωνική πρόνοια. Αυτό είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει σε άλλες εκθέσεις με άλλα θέματα και σε σχέση με το ποιο θα είναι το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Θέλουμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά να ληφθούν υπόψη, κυρίω για να καλυφθούν οι δραστηριότητε τη ερασιτεχνική αλεία, ο ρόλο των γυναικών στι παράκτητε περιοχέ και η ε, καλή διεξαγωγή ενός κοινωνικού διαλόγου. Και επίσης είναι σημαντικό πάνω απ' όλα η Επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη να διαχωρίζει τη θέση της ε, σε σχέση με το τι θέλει να γίνει για τις επενδύσεις των παράπλευρων δραστηριοτήτων της ερασιτεχνικής αλίας και των ειδικών τοπικών δραστηριοτήτων συμμετοχικού χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή έχουν, υπάρχει, υπάρχουν υποδομές που έχουν εγκαταλειφθεί ε, γιατί δεν χρησιμοποιούνται πλέον, μπορούν όμως να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει. Θα μπορούσαμε να προβλέψουμε δημοσιονομικές γραμμές για το σκοπό αυτό, διότι μόνο με μια πολιτική συνεργασία και κοινή διαχείριση των ηχθικών πόρων ε, θα μπορέσουν θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή αποκατάσταση των αποθεμάτων και την καλή λειτουργία της πολιτικής αλίας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Φίτο, έχετε και εσείς το λόγο ως σκιώδης. Παρακαλώ να είστε και εσείς σύντομος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Πρόεδρε, τρία πράγματα. Ξεκινώντας από την καλή βάση ε, για την πρόταση, από τις της εισηγήτριας, εδώ να αναπτύξουμε τρία θέματα. Η γραμμή της απλούστευσης που προβλέπεται και από τους άλλους κανονισμούς. Οι επιχειρηματίες του χώρου πρέπει να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα εργαλεία με συμμετοχή και καλή διοργάνωση της επαγγελματική τους ε, κατηγορίας. Επίσης, η δράση που θα, εφαρμο... θα προβλεφθεί πρέπει να επιτρέψει να αντιμετωπιστούν και οι έκτακτες συνθήκες, κλιματικές και περιβαλλοντικές, με μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός ταμείου εγγύησεων για τους αλληλείς. Τρίτο σημείο, ο κοινωνικονομικός ρόλος των δραστηριοτήτων του όλου τομέα με κίνητρα για μέτρα που θα στηρίξουν τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την αλία και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Αυτά είναι τα θέματα για τα οποία θέλουμε να υποβάλουμε τροπολογίες. Πιο γρήγορα δεν μπορούσα να τα πω. Thank you. Uh, ε, ευχαριστώ. Εγώ είμαι σκιώδης ηγητρία σε αυτήν την Επιτροπή, αλλά και στην Επιτροπή Αλίας. Και συμφωνώ με το όραμα των συναδελφών, ειδικά του κυρίου Ομαζή η πρόταση της Κομισιόν σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, αλλά δυστυχώς δεν σέβεται της αρχή της αναλογικότητας. Η πρόταση πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλα τα κράτη-μέλη από πλευράς αλλιευτικών περιοχών, γιατί σε κάποιες περιοχές η παράκτια αλληλεία μικρής κλίμακα είναι μη βιώσιμη και θεωρώ ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε τις αλληλευτικές δυνατότητες. Όσον αφορά το Ταμείο έχουμε υποβάλει πολλές ε, τροπολογίες για ευελιξία και απλοποίηση. Θεωρούμε ε, πολύ σημαντική την υδατοκαλλιέργεια ε, ως εναλλακτική στην εμπορική αλία που θα μειώσει τις πιέσεις στα ίχθη αποθέματα και το στηρίσμα, όσον αφορά και το ποσοστό συγχρηματοδότησης που θεωρούμε ότι πρέπει να αυξηθεί. Και τέλος, το ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάποιες δράσεις πρέπει να αυξηθεί, να στηρίξουμε τις καινοτόμες δράσεις στο τοπικό επίπεδο, να προωθήσουμε την ε, τοπική στρατηγική ανάπτυξης, ε, νέους ψαράδες, ε, προστασία της βιοπικιλότητας, διαφοροποίηση του εισοδήματος, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες αποζημιώσεις ε, όταν σταματάει προσωρινά η αλληλεία. Όλα αυτά θεωρώ ότι μπορεί να δώσουν προσθέμενη αξία στον τομέα αλληλείας και χθεοκαλλιέργειας. Θα προωθήσω το όραμά σας. Ε, οι τροπολογίες μου πάνε στην ίδια γραμμή και ελπίζω στο μέλλον να συνεχίσει το Ταμείο να λειτουργεί εύρυθμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Νταμάτο, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τα θέματα του περιβάλλοντος συμφωνούμε και θα υποβάλουμε σχετικώς τροπολογίες για να στηρίξουμε τα, της βιωσιμότητας, γιατί θέλουμε να ενισχυθεί και το άρθρο της βιολογικής και της κοινωνικής βιωσιμότητας ταυτόχρονα. Προσοχή στο άρθρο 14, ως προς τις διατάξεις για την ανάπτυξη της μικρής αεραστεχνικής αλίας, θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση της πιστώσεως και στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, στην παράγραφο 17, στο άρθρο 17, με μια τροπολογία που θα επιτρέψει να υπάρξει ανανέωση στι γενιέ των αλλιέων και με τη χρήση νέων σκαφών, τα οποία όμω δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την συνολική δυνατότητα αλλίευση. Ε, το Ταμείο θα πρέπει να επιτρέπει να προβλεφτούν δράσει για την κατάρτιση και την εκπαίδευση των νέων, να υπάρχει επαγγελματική επικαιροποίηση των γνώσεων των αλλιέων για την προστασία του περιβάλλοντο και την ε, βιοπικιλότητα, ε, την ασφάλεια τη ζωή στη θάλασσα και την ασφάλεια των εργαζομένων στα αλληλευτικά σκάφη. Επίση, το άρθρο 17, και εδώ θα ολοκληρώσω, πρέπει να προβλέψουμε ένα νέο εδάφιο, το οποίο να αποσαφηνίζει πώ το, το Ταμείο θα επιτρέπει την πρόσβαση επιχειρήσεων τη υδατοκαλλιέργεια σε εργαλεία διαχείριση των κινδύνων, με τη κίνητρα για τις πολιτικές ασφάλειες της και ε, τη Θα πρέπει να μπορούν να καλύπτονται οι απώλειε που οφείλονται σε κλιματικέ ε, καταστροφέ ε, περιβαλλοντικές και το τι θα γίνεται για τους αλλοί σε περίπτωση ατυχήματος στη θάλασσα κατά την εξαγωγή της δουλειά τους. Τώρα δίνω τον λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομη, σας το υπόσχομαι. Επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα σχόλια. Θα ήθελα να εστιάσω σε δύο-τρία. Το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω είναι η απλοποίηση της υλοποίησης και έχουμε έτσι ένα ευρύ φάσμα επιλέξιμων ε, δράσεων. Το ότι δεν έχουμε έναν αναλυτικό κατάλογο σημαίνει ότι μπορούμε να στηρίξουμε τα πάντα μέσω του Ταμείου, εκτός βεβαίως από ε, τον ξεκάθαρο κατάλογο μη επιλέξιμων ε, δράσεων. Θεωρούμε ότι έτσι έχουν τα κράτη-μέλη την ευελιξία που απαιτείται για να προσαρμόσουν τη στήριξη στις ανάγκες τους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όλοι οι τομείς στήριξης ε, που αναφέρατε σήμερα, όπως ο ρόλος των γυναικών, η κατάρτιση, όλα αυτά είναι ήδη επιλέξιμα. Ο δεύτερος στόχος που θα ήθελα να αναφέρω είναι η ότι η νέα αυτή πρόταση έχει στόχο να στοχεύσει καλύτερα στην επιτευξή των στόχων της ε, κοινή ε, αλληλευτικής πολιτικής. Ε, να συμπενθυμίσω το ταμείο αυτό είναι το Κοινοτικό Ταμείο Αλίας, οπότε καλύπτει βεβαίως τους στόχους κοινή αλληλευτικής πολιτικής, αλλά και την βιώσιμη ηχθειοκαλλιέργεια την προώθηση θαλασσίων οικοστημάτων, τη γαλάζια οικονομία, τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά την διαχείριση των ωκεανών. Αλλά το ΠΔΠ είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό σε τοπικό επίπεδο. στις παράκτιες ε, κοινότητες ε, μέσω της στήριξης που υπάρχει για το θέμα αυτό. Ένα σχόλιο τώρα για το δημοσιονομικό πλαίσιο προτείνουμε μια μείωση 5% που ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις συνέπειες ε, του Brexit στον προϋπολογισμό. Ο υπολογισμός μας δείχνει ότι τα κράτη-μέλη σε ονομαστικούς όρους ε, θα διατηρήσουν 96,5% των τρεχόντων φακέλων. Τέλος, μια κουβέντα για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Σε σχέση με αυτές ε, πιστεύουμε ότι το μελλοντικό ταμείο ε, φροντίζει επαρκώς ε, τις ανάγκες αυτών των περιεχών. Οπότε η Κομισιόν πρότεινε μια νέα στρατηγική ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις απομακρυσμένες περιοχές που βασίζεται σε σχέδια δράσης με δεσμευμένα ποσά μέχρι και 50% των ποσών αυτών καλύπτουν ε, το επιπλέον κόστος ως αποζημίωση. Το υπόλοιπο θα πρέπει να στηρίζει διαρθρωτικές επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία και την αλία επιπλέον. Προβλέπεται ένα υψηλότερο ποσοστό ε, συγχρηματοδότηση, 85% αντί για 50% για τις εξόχως μακρισμένες περιοχές. Αυτό μαζί με την ε, προτιμησιακή μεταχείριση που προτείνουμε για τις μικρές αληφτικές ε, παράκτιες ε, μονάδες ε, θα δώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε οι περιοχές αυτές να αναπτυχθούν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ομαρζέ. Μπορείτε να ολοκληρώσετε την συζήτηση σύντομα κι εσείς. Ναι, θα προσπαθήσω να απαντήσω γιατί ψηφίζουμε στις δύο, αλλά από όλε τις παρεμβάσεις βλέπουμε ότι συγκλίνουν οι θέσει όλων των μελών τη Επιτροπή. Δεν νομίζω θα είναι δύσκολο να έχουμε μια θέση που να εκφράζει όλου. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σύντομο. Πολύ ευχαριστώ. Και τώρα θα παρακαλέσω τους συντονιστές να παραμείνουν. Αχ, με συγχωρείτε, το ξέχασα. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών της νομοδότησης αυτής 5η 8 Νοεμβρίου. Το μεσημέρι στις 12. 8 Νοεμβρίου 5η. Διάφορα, δεν έχουμε χρόνο για διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση 15 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. 10 λεπτά για τους συντονιστές. And we have only actually one issue. Ένα θέμα έχουμε εδώ Εάν μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις συνεδρίες των συντονιστών, αμέσως. Ένα μόνο θέμα